Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνεδρίασή μας. Στην αρχή της συνεδρίας αυτής θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα ασκουμένων από την Πράγα, από την ε, ανώτατη ε, σχολή Διοίκηση ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν έρθει για να δούνε πώς λειτουργεί η Επιτροπή μας. Περάσουμε στο πρώτο σημείο της μερίσιας διάταξης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προτείνω τις ακόλουθες αλλαγές. Τα σημεία 15, 16, 18, 29 και 30 αναβάλλονται και το σημείο 31 σας προτείνω να εξετάσουμε μετά το σημείο 28. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Συνεπώς εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Τώρα σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Να σας μερώσω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου και των Στονιστών της Επιτροπής μας στις 2 Οκτωβρίου. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι ο κύριος Λεμπρετών θα διοριστεί ως εισηγητής για την υπεράσπιση των προνομίων και αλυσιών της κυρίας Ελεονόρα Φορέντσα. Ο κύριος Χρυσόγονος έχει διοριστεί ε, εισηγητής όσον αφορά την έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του ενωσιακού δικαίου, ετήσια έκθεση του 2016. Και ο υποφαινόμενος θα συνυπογράψει μια κοινή επιστολή των Προέδρων Γιούρι και Λίμπε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά τον εξορθολογισμό μέσων και εργαλείων πολιτικής του νοσιακού αστικού δικαίου και του δικαίου περιασύλου σε σχέση με τη μετανάστευση. Αυτά όσον αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών. Σημείο 3 τώρα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση των πρακτικών υποβληθούν ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θεωρείται ότι ε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 19 και 20 Ιουνίου, 12 και 13 Ιουλίου και 7 Σεπτεμβρίου εγκρίνονται. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε τις έκθεσεις EPRS σχετικά με τις αιτήσει επιστροφής έργων τέχνης που ληλατήθηκαν. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τον καθηγητή κύριο Ματίας Βέλερ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την μελέτη του όσον αφορά την ε, διασυνοριακή υποβολή ετοιμάτων επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο λιλασίας σε ένοπλες συγκρούσεις σε πολέμους. Θα δώσω όμως ε, τον λόγο στον κύριο Βέλερ τώρα. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τα βασικότερα πορίσματα της μελέτης αυτής όσον αφορά τις αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης που λιλατήθηκαν και σχετικών πολιτιστικών αγαθών σε σχέση με την πιθανή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαμε να είχαμε μέσω ενωσιακή νομοθεσίας για το ζήτημα αυτό. Να ξεκινήσω καταρχάς με μία σύντομη εισαγωγή για τη μελέτη αυτή. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα δηλαδή αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Προσπαθήσαμε να θέσουμε αυτό ως βάση. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε καταρχάς ότι υπάρχει παράνομο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα, μολονότι ακόμα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα για, την, για το εύρος του φαινομένου αυτού. Γιατί συνειδητοποιείται ότι το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με, την, με εγκληματικές δραστηριότητες, με την παράνομη παράτυπη αγορά, επομένως δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα και επίσημα αριθμητικά δεδομένα. Εμέσω πάντω υπάρχουν διάφορα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θεωρούμε ότι υπάρχει όντω ένα σημαντικό πρόβλημα και ότι γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να ανησυχούμε. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε εκθέσεις της Interpol ή ακόμα και σε εκθέσεις του FBI για το ζήτημα αυτό ή ακόμα και σε πρόσφατα μέτρα που έχει λάβει το Συμβούλιο της Ευρώπης ή θα μπορούσαμε ακόμα και αναφερθούμε σε εκθέσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες αυτές οι εκθέσεις αναφέρονται στο πρόβλημα αυτό και στο γεγονός ότι ε, οι τρομοκρατικές οργανώσεις όλο και περισσότερο προσπαθούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του εμπορίου λιλατημένων έργων τέχνης. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν μέχρι ενός βαθμού συνδέονται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δημόσιο δίκαιο και ξέρετε το ζήτημα αυτό είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και γνωρίζουμε και από άλλες προβληματικούς τομεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση ενός τόσο δύσκολου προβλήματος είναι να χρησιμοποιήσουμε μέτρα του δημοσίου και του ιδιωτικού δικαίου. Το δεύτερο πόρισμα λοιπόν της μελέτης μου θα ήταν να προτείνω την ακόλουθη προσέγγιση, συνδυασμός μέτρων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Χρειαζόμαστε δηλαδή τόσο ιδιωτική όσο και δημόσια επιβολή μέτρων. Από την πλευρά του δημοσίου δικαίου έχουμε πολύ περισσότερα μέτρα. Θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στον τομέα του ιδιωτικού δικαίου και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για ιδιωτική επιβολή. Τώρα τι εννοούμε λέγοντας ιδιωτική επιβολή. Η ιδιωτική επιβολή βασίζεται κυρίως σε αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του αστικού δικαίου και που έχουν να κάνουν με την επιστροφή έργων τέχνης. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα τρία βασικότερα πορίσματα όσον αφορά την κατάσταση όπως έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Βάσει της τρέχουσας λοιπόν αυτής υφιστάμενης κατάστασης, θα ήθελα να σας προτείνω τις ακόλουθες συστάσεις. Στόχος των συστάσεων αυτών είναι να βελτιωθεί το σύστημα αστικού δικαίου, το σύστημα υποβολής αιτήσεων μέσω του αστικού δικαίου όσον αφορά τα έργα τέχνης που έχουν ληλατηθεί και γενικότερα τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν λελατηθεί. Όσον αφορά τώρα το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή δικαιοδοσία, το ζήτημα το οποίο τίθεται συνήθω είναι ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο και σε ποια χώρα κάθε φορά που υπάρχει μία υπόθεση δικαστική που έχει πολλές διεθνεί πτυχές. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα μέσο αυτή τη στιγμή. Είναι ο κανονισμός 1α των Βρυξελών του 2012. Θα έλεγα ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχείς ε, κανονισμούς που έχουμε στα πλαίσια του νησιακού δικαίου όσον αφορά για τις δικαστικές αυτές υποθέσεις και στην επαναδιατύπωσή του προβλέπεται πλέον μια νέα διάταξη για την αποκατάσταση έργων τέχνης που έχουν λελατηθεί, άρθρο 7 σημείο 4. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα όσον αφορά το άρθρο, το, το άρθρο αυτό, το θα έπρεπε καταρχά να παληφθούν τα τεχνικά αυτά προβλήματα προτού χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό για τα ζητήματα αυτά δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή. Μπορώ πάντω να σα δώσω, αν το επιθυμείτε, περισσότερε πληροφορίε στη συνέχεια για τα τεχνικά αυτά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει σε σχέση με το άρθρο 7.4 του κανονισμού αυτού. Ένα άλλο σημείο τώρα που ενδεχομένω να μην συνδέεται άμεσα με το δικό μα το ζήτημα έχει να κάνει με την ασυλία που προβλέπεται κάθε φορά που ένα κράτος μέλος έχει δανείσει ένα εργοτέχνης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και αν στην περίπτωση αυτή τίθεται ένα ζήτημα επιστροφής του συγκεκριμένου αυτού έργου τέχνης σε κάποια άλλη χώρα. Ξέρετε ότι ε, προκύπτει το ζήτημα αυτό πολύ συχνά σε περιπτώσει δανεισμού έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών από το ένα κράτο μέλος στο άλλο. Ορισμένα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν ένα καθεστώς κατά της κατάσχεσης, αλλά κράτη-μέλη δεν έχουν τέτοια νομοθεσία και όποτε υπάρχει ένα τέτοιο καθεστώς κατά της κατάσχεσης του την ένωμη τάξη ενός κράτους μέλους, τότε στην περίπτωση αυτή προκύπτει ένα πρόβλημα για τον ετούντα, την επιστροφή του εργοτέχνης. Από την άλλη, μην ξεχνάμε όμως ότι το προστατευτικό αυτό καθεστώς κατά της κατάσχεσης τουλάχιστον δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης κυκλοφορίας των έργων τέχνης μεταξύ των κρατών μελών και προωθούν αυτό το οποίο ονομάζουμε δημόσια πρόσβαση στον πολιτισμό, στα πολιτιστικά αγαθά και αυτό το οποίο αποκαλούμε κινητικότητα των συλλογών έργων τέχνης. αυτό το καταστατικό, αυτά τα μέτρα κατά της κατάσχεσης θα πρέπει να ισορροπηθούν εκεί πέρα που υπάρχουν με τα συμφέροντα των ιδιωτών όσων δηλαδή υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή τέχνης και θα πρέπει να υπάρχει εν συνεχεία μια εναρμόνιση του καθεστώτος αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία 2014-60, όσον αφορά την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παρανόμως απομακρυνθεί από την επικράτεια ενός κράτους μέλους. Η οδηγία αυτή ακόμα δεν ασχολείται με το ζήτημα της ε, ασυλίας, αλλά θα μπορούσαμε να μεταρρυθμίσουμε την ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιώντας την οδηγία αυτή, την οδηγία 60 του 2014. Ένα τρίτο σημείο τώρα, η επιλογή του δικαίου. Κάθε φορά που προκύπτει μία σύγκρουση με άλλες δικαιοδοσίες, με άλλα ένομα συστήματα, τίθεται το εξή ερώτημα. Ποιο είναι το ουσιαστικό δίκαιο το οποίο θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση αυτή. Θα είμαι πολύ σύντομος για το σημείο αυτό. Έχει γίνει ήδη μια εκτενέστατη συζήτηση στα πλαίσια των ενδιαφερομένων για το ζήτημα αυτό, των ομομαθών, στα πλαίσια του ιδιωτικού και του διεθνούς δικαίου και πολλοί προτείνουν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία, ένα ενιαίο δίκαιο προκειμένου να προστατεύονται αυτά τα πολιτιστικά αγαθά. Στο, στη Βελγική, για παράδειγμα, νομοθεσία υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα και η πρότασή μου θα ήταν να εναρμονιστεί αυτή η δυνατότητα επιλογής δικαίου όσον αφορά τα έργα τέχνης και τα πολιτιστικά αγαθά, ακολουθώντας ή ευθυγραμμιζόμενη με την βελγική νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα το ουσιαστικό δίκαιο, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η νομοθεσία για την απόκτηση καλή την πίστη, καθώς επίσης και η νομοθεσία όσον αφορά την περιοριστική απόκτηση πολιτικών αγαθών, πάντα χρησιμοποιείται στα πλαίσια του αστικού δικαίου κάθε φορά που υπάρχει μια διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Εδώ πέρα όμω διαφέρουν πάρα πολλοί σχετικέ νομοθεσίε των κρατών μελών. Παράλληλα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε νομοθεσία υιοθετείται αναδρομικά, ουσιαστικά δεν θα πρέπει να ισχύει, δεν μπορεί να ισχύει στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεδομένων λοιπόν των δύο αυτών σημείων, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε μια κάποια πρόοδο στο σημείο αυτό, αν θα ρίναμε τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση στην σύμβαση UNIDROIT του 1995, μια σύμβαση στην οποία ήδη έχουν προσχωρήσει ως συμβαλόμενα μέρη ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά πάλι όχι. Η σύμβαση αυτή έχει να κάνει πάλι με ζητήματα ιδιωτικού δικαίου όσον αφορά την καλή τυπίστη απόκτηση πολιστικών αγαθών και ασχολείται και με κάποια άλλα παρεμφερή ζητήματα. Αν προσχωρούσαν λοιπόν τα κράτη-μέλη στη σύμβαση αυτή, θα μπορούσαμε όντω να επιλύσουμε πολλά ζητήματα. Από την άλλη θα μπορούσαμε να ενσωματώναμε ένα τμήμα της σύμβασης αυτής ως μέσο παράγωγου ενωσιακού δικαίου και αυτό θα μπορούσε να γίνει ως εξής. Θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε το ουσιαστικό ιδιωτικό δίκαιο της σύμβασης αυτής στην οδηγία 60 του 2014 την οδηγία δηλαδή αυτή που αναφέραμε πριν από λίγο σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Μία τρίτη πιθανότητα θα ήταν να ενσωματώναμε τους κανόνες για την καλή την πίστη απόκτηση των πολιστικών αγαθών από το σχέδιο πλαισίου αναφοράς πάλι στην οδηγία αυτή Και με τις δύο αυτές λοιπόν πιθανές προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση θα βελτιώναμε το ένομο καθεστώ Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε ένα ιδιαίτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τα έργα τέχνη που έχουν λαιλατηθεί από του Ναζί. Πάλι εδώ πέρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε νομοθεσία με αναδρομική ισχύ δεν μπορεί να γίνει δεκτή στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χάρτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμείς να νομοθετήσουμε με αναδρομική ισχύ σε σχέση με συναλλαγές που λάβανε χώρα στο παρελθόν και που μετέφεραν την κυριότητα έργων τέχνης από το ένα άτομο στο άλλο, αν η συναλλαγή αυτή θεωρεί το ένομη την εποχή εκείνη και έγκυρη την εποχή που έγινε εκείνη η συναλλαγή. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να βελτιώσουμε την ένομη κατάσταση όσον αφορά το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε διαφορετικές πάλι προσεγγίσεις ή πιθανές λύσεις. Εμείς στη μελέτη μας προτείνουμε δύο πιθανούς τρόπους για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε την εν λόγω κατάσταση σε σχέση με αυτά τα έργα τέχνης τα οποία λατήθηκαν από τους Ναζί. Μία πιθανότητα θα ήταν να τροποποιηθεί το δίκαιο που διέπει τις συνθήκες εμπορίου για τις μελλοντικέ συναλλαγές, το εμπορικό δηλαδή δίκαιο, και θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε μια νέα νομοθεσία, δημιουργώντας μια οδηγία, για παράδειγμα, που θα έχει να κάνει με την πώληση συγκεκριμένων πολιτιστικών αγαθών που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των έργων τέχνης που έχουν λελατηθεί από τους Ναζί. Μια άλλη πιθανότητα θα ήταν να προβλεφθούν συγκεκριμένα ένδικα μέσα για τον πολιτή, όσον αφορά την, συγγνώμη, τον αγοραστή, όσον αφορά την προέλευση των έργων τέχνης που του προτείνει ο πολιτής. Στην περίπτωση αυτή θα διασφαλίζαμε ότι τα συμβαλόμενα μέρη στα πλαίσια μιας σύμβασης αγοράς και πώλησης θα γνωρίζανε και τα δύο τελικά τι πωλείται και θα γνωρίζανε αμέσως ότι η πώληση μπορεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση να έχει να κάνει με ένα έργο τέχνης που έχει λαιτηθεί από τους Ναζί. Στην περίπτωση αυτή η τιμή του προϊόντος θα μπορούσε να υποτιμηθεί πολύ σημαντικά γιατί ουσιαστικά κανείς δεν θα ήθελε να αγοράσει ένα έργο τέχνης το οποίο αποτελεί αντικείμενο λελασία από τους Ναζί. Θα μπορούσε η διάσταση αυτή να αποτελέσει πτυχή του εμπορικού δικαίου που θα διέπει τέτοιε αγοραπολισίε και που θα επιτρέπει στα δύο συμβαλόμενα μέρη να γνωρίζουν τελικά τι πολλούν και τι αγοράζουν. Θα μπορούσαμε επίση να βελτιώναμε τι λύσει που προβλέπονται πέρα από το ίδιο το δίκαιο. Ακριβώ επειδή υπάρχουν συγκεκριμένε δυσκολίε στα πλαίσια του αστικού δικαίου κυρίω, 44 κράτη αποφάσισαν το, αποφάσισαν το 1998 να χρησιμοποιήσουν μία μορφή ήπιας νομοθεσίας τις αρχές της Ουάσιγκτον, δηλαδή όσον αφορά τα έργα τέχνη που λατήθηκαν από τους Ναζί. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, στόχος μας είναι σε κάθε περίπτωση να μπορούμε να βρίσκουμε δίκαιες λύσεις για την αποκατάσταση αυτών των έργων τέχνης ή τουλάχιστον για να ληφθεί υπόψη ότι τα συγκεκριμένα αυτά έργα τέχνης εμπίπνε στην κατηγορία των πολιτιστικών εκείνων αγαθών που έχουν ελληλατηθεί από τους Ναζί. Υπάρχουν επίσης και συγκεκριμένες συστάσεις από κράτη-μέλη όπως οι κάτω χώρες, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία και οι φορεί που έχουν προτείνει συστάσει στι χώρε αυτέ προσπαθούν να βρουν πάλι δίκαιε λύσει για προβληματικέ υποθέσει προσπαθούν επίσης από δεντολογικής πλευράς να προτείνουν συγκεκριμένες δίκαιες ε, ισότιμες λύσεις. Ένα σημαντικό λοιπόν μέτρο θα ήταν να επαναλάβουμε κάποιες βασικές αρχές βάσει των οποίων μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τέτοιες υποθέσεις. Πώς μπορούμε δηλαδή να εφαρμόσουμε καλύτερα τις διοντολογικές αρχές, τις αρχές ηθικής που αποτελούν ουσιαστικά βάση των συστάσεων αυτών που έχουν υποβάλει, όπω σας είπα, διάφορα κράτη-μέλη. Περνώ στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασή μου στο οποίο θα ήθελα να σας δώσω, να σας προτείνω κάποια συμπληρωματικά μέτρα, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τα μέτρα αυτά τα οποία σας πρότεινα πριν από λίγο. Ένα πρώτο τέτοιο μέτρο θα ήταν να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την έρευνα της διασυνοριακής προέλευσης πολιτιστικών αγαθών, έχοντας βάσεις δεδομένων με μεταδεδομένα, όπου θα συλλέγουμε δεδομένα από τα κράτη-μέλη, θα τα ομαδοποιούμε και θα τα διατίθουμε έπειτα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σαφές ότι όλη η έρευνα που γίνεται σε σχέση με την προέλευση ενός πολιτιστικού αγαθού είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και ιδιαίτερα ακριβή, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά που υπάρχει κάπου μια πληροφορία για την προέλευση ενός πολιτιστικού αγαθού, η πληροφορία αυτή να γίνεται άμεσα διαθέσιμη σε όλους. Κάτι ότι δεν συμβαίνει ακόμα και αν είχαμε μια τέτοια κεντρική βάση δεδομένων θα βελτιώναμε πάρα πολύ την κατάσταση. Σε σχέση με αυτό θα πρέπει να έχουμε και ένα κοινό σύστημα απαρίθμησης ε, για τα πολιτιστικά αυτά αγαθά και να έχουμε τελικά έναν κοινό κατάλογο όπου θα μπορούμε τελικά να συμπεριλαμβάνουμε όλα αυτά τα πολιτιστικά αγαθά και ιδίω τα πολιτιστικά εκείνα αγαθά τα οποία είναι τα πιο επίμαχα, αν θέλετε. Αυτά τα οποία ενδεχομένω μπορούν να αποτελούν αντικείμενο λιλασίε από του Ναζί. Θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο, έχοντα τον κατάλογο αυτό και έχοντα και ένα κωδικό που θα συνοδεύει τα προϊόντα, να γνωρίσουμε τελικά ποια είναι τα προϊόντα αυτά, ποιο τα αγοράζει και ποιο τα πουλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε επίση και εναλλακτικού τρόπου επίλυση διαφορών Ξέρετε ότι το σύστημα αυτό προβλέπεται σε άλλους τομείς δικαίου, αλλά δεν έχουν καταβληθεί ακόμα πάρα πολλές προσπάθειες προκειμένου να ισχύουν εναλλακτικέ μορφές επίλυσης διαφορών στον τομέα των έργων τέχνης που έχουν ελελατηθεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν φορέα που θα μπορούσε τελικά να συμβάλλει σε αυτή την εναλλακτική επίλυση δικαστικών διαφορών. Τέλος, σε βάθος χρόνου νομίζω ότι θα πρέπει ενδεχομένω να δημιουργήσουμε και έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, η οποία υπηρεσία θα μπορούσε να μαδοποιήσει αν θέλετε όλα αυτά τα μέτρα. Στην τελευταία αυτή διαφάνεια θα ήθελα να συνοψίσω την λεγόμενη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των μέτρων αυτών. Θα να καταρχά ότι τα τρία πρώτα ζητήματα, η δικαιοδοσία, η ασυλία και η επιλογή δικαίου, συμβάλλουν σαφώ να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αλλά βέβαια είναι ζητήματα που έχουν κυρίω τεχνική φύση και επομένω έχουν ε, περιορισμένη αν θέλετε αποτελεσματικότητα στην πράξη. Θα επέπεινε λοιπόν περισσότερο στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη πρόταση που σας έκανα, που έχει να κάνει με το ουσιαστικό δίκαιο και ιδίω ε, με τις προτάσεις που σας έκανα για την καλή πίστη απόκτηση πολιτιστικών αγαθών, τι προτάσει που γίνανε όσον αφορά την ειδική αντιμετώπιση των εργοτέχνης που έχουν τεθεί από του Ναζί και η έκτη πρόταση που έχει να κάνει με τα συμπληρωματικά αυτά μέτρα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τα μέτρα τα οποία σα παρουσίασα στην αρχή. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι προφανώς διαθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Λέει ο Πριν να δώσουμε τον λόγο για ερωτήσεις και απαντήσεις να δώσω τον λόγο στον κύριο Κρίστιανσον του EPRS που θα συνεχίσει από εκεί που το αφήσατε εσείς το θέμα για την αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δική μου συνεισφορά είχε μάλλον τον στόχο να κάνει την εισαγωγή για τη μελέτη του καθηγητού. Να βάλω το πλαίσιο δηλαδή και μετά να του παραδώσω το μικρόφωνο για να αναπτύξει τα βασικά θέματα τα οποία ήδη έκανε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Άρα, λέει ο Πρόεδρος, μπορούμε να περάσουμε μέσω της ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεν βλέπω κανένα να γύρει ενδιαφέρον. Εγώ βεβαίως έχω μια ερώτηση. Α, εσείς κύριε Φως, έχετε ερώτηση. Έχετε βεβαίως προτεραιότητα απέναντί μου. Πρώτα ευχαριστώ εγκάρδια τον κύριο καθηγητή. Λόγω προηγούμενων υποχρεώσεων δεν πρόλαβα να τα ακούσα όλα. Όμως, εάν συγκρίνετε τις προτάσεις σας με τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί η λαϊλασία έργων τέχνης στη Γερμανία, υπάρχει ένα σύστημα καταχώρησης σε μητρώα αγνοωμένων καλλιτεχνημάτων. Το ζήτημα της ιδιότητας του κυρίου μετά από τόσα πολλά χρόνια που έχουν περάσει και πράγματα τα έχουν χάθει και ούτω καθεξής, θεωρείτε ότι είναι συγκρίσιμο το καθεστώς αυτό με τα όσα προτείνεται ή πού βλέπετε να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές και τι θα συστήνατε σε μια χώρα όπως η Γερμανία σε ό,τι αφορά την βελτίωση του καθεστώτος αυτού. Γιατί για μένα αυτό είναι λίγο πολύ το state of the play. Δεν έχω εικόνα για τα άλλα νομοθετήματα που παίζουν εδώ ένα ρόλο, δηλαδή σε άλλες χώρες. Αλλά σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, ας το πω έτσι. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες. Ε, κινώντα από την βάση που έχουμε ήδη στη θέση μας. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας, απαντά ο καθηγητής Μίλλερ, και βεβαίω θα απαντήσω στα γερμανικά, μια και με ρωτήσατε στα γερμανικά. Αναφέρεστε στα λατημένα καλλιτεχνήματα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό στην Γερμανία. Και λέτε επίση ότι η Γερμανία έχει καταβάλει πολύ άριθμες προσπάθειες ήδη να δείξει προοδευτική ε, προσέγγιση και να δει τι μπορεί να κάνει για να αποζημιώσει κιόλα τα πρόσωπα αυτά που έχουν δεινοπαθεί στο παρελθόν. Πράγματι έχουν ληφθεί πολλά μέτρα από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση. Υπάρχει και στο Μαγδεμβούργο κέντρο, ίδρυμα δηλαδή το οποίο χρηματοδοτούν τα ομόσπονδα κρατήδια για να ε, εγκύπτει στα θέματα αυτά, να εγγράφονται τα καλλιτεχνήματα, τα διάφορα καλλιτεχνικά έργα σε τράπεζες δεδομένων η εμπειρία όμως από τις τράπεζες αυτές δεδομένων είναι ότι η καταχώρηση στοιχείων προελεύσεως, δηλαδή ποια ήταν η μοίρα του καλλιτεχνήματος τότε και τι έχει γίνει στην πορεία μέχρι τώρα, είναι ιδιαίτερα δαπανηρά και χρονοβόρα. Έχει λοιπόν έρθει, θεωρώ, η χρονική στιγμή όπου τα συλλεγόμενα δεδομένα από τα μουσεία όπου γίνονται έρευνες να συγκεντρωθούν, να συλλεχθούν και να συγκεντρωθούν. Πρώτα-πρώτα σε επίπεδο Ομοσπονδιακής Γερμανίας και για την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Σε ένα δεύτερο βήμα, αυτό που ανέφερα εγώ προηγουμένως ως συμπληρωματικά μέτρα, που θα είναι ένα σημαντικό βήμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να συγκεντρωθούν δηλαδή τα δεδομένα αυτά σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο για να απλοποιηθεί η διαδικασία διαπίστωσης της προέλευσης και χρειάζονται μεγάλε προσπάθειε. Αλλά αυτή είναι η διασύνδεση που βλέπω ανάμεσα στι προσπάθειε που καταβάλλονται τώρα στη Γερμανία και τι ενδεχόμενε βελτιώσει που θα μπορούσαν να επισυμβούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Μπερζερόν. Γνωρίζω το γαλλικό δίκαιο, λιγότερο το ευρωπαϊκό. Στο γαλλικό δίκαιο αυτός που αποκτά καλή την πίστη, χρωστά το τίμημα και όχι το αντικείμενο. Στο γαλλικό δίκαιο αγοράζεται σε μια δημοπρασία ένα ε, παλαιό ορολόγιο, διαπιστώνεται ότι είναι κλιμαίο, δεν αποδίδεται το ρολόι, αποδίδεται το τίμημα που πληρώσατε. Για μένα αυτό είναι κάτι το ε, απίστευτο. Και βεβαίω η ιστορία με τα κλοπημένα των Ναζί είναι ε, γνωστή και συνταρακτική. Αλλά υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο ε, με ανησυχεί πάρα πολύ, με ανησυχούσε και με ανησυχεί, ο αριθμός ε, αντικειμένων αφρικανικής προελεύσεως που πολλούνται σε διεθνείς αγορές και που ίσως να μην έχουν μεγάλη εμπορική αξία, έχουν όμως πολιτιστική αξία και πολιτισμική και ηθική αξία πάρα πολύ σημαντικές. Παράδειγμα, προσωπικής εμπειρίας. Αγόρασα ένα αντικείμενο αφρικανικής τέχνης. Το αγόρασα, ήταν μια κεφαλή μέσα σε ένα σάκο οστών. Και έψαξα και βρήκα ότι το αντικείμενο αυτό κανονικά δεν εγκαταλείπει ποτέ το σπιτικό του Αφρικανού κυρίου, διότι εκπροσωπεί όλους τους προγόνους, όλης της οικογένειας. Και ο αρχηγός της οικογένειας κοιμάται έχοντας αυτό το αντικείμενο δίπλα του. Πώς είναι δυνατόν το αντικείμενο αυτό να καταλήξει σε μια δημοπρασία, σε δημόσια πώληση και εγώ να το αποκτήσω, να γίνω κυρία. Βλέπω εδώ να υπάρχει μια πτυχή της ζωής του δυτικού ανθρώπου, η οποία δεν θα τον κάνει υπερήφανο. Σαν να πουλάν όλα τα ε, ιερά κοιμήλια των Ευρωπαίων στην Αφρικανική αγορά. Διότι δεν αποδίδουμε την ίδια αξία που αποδίδουν οι Αφρικανοί. Είναι σχεδόν και ανθρωπολογικό πρόβλημα αυτό, διότι δεν δίνει κανείς στους άλλους μια αξία εσωτερική που έχουν τα αντικείμενα. Διερωτώ με, εάν το κείμενο που ε, συντάσσεται τώρα και που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως θα πρέπει να λάβει υπόψη και την πτυχή αυτή. Διότι αυτά πάμε και κλέβουμε από τους άλλους. Και για τους Λατινοαμερικανούς, με όλα τα πρεκολομβιανά αντικείμενα που δεν επιτρέπεται πλέον η πώλησή τους, χωρίς να περιγράφεται ακριβώς η προέλευσή τους. Είναι σημαντικό να επεκταθεί η διάσταση αυτή του διεθνούς δικαίου και στους Αφρικανούς. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πολύ σημαντική ε, ερώτηση. Δείξατε πολλά σημαντικά σημεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρώτο. Έγινε ακόμη πιο σαφές ότι υπάρχουν ε, ουσιαστικές διαφορές στην νομοθεσία περί της απόκτησης καλή στη μεταξύ των κρατών μελών. Δεν υπάρχει μια τέτοια ευρωπαϊκή νομοθεσία ακόμη και ακριβώς ε, σε αυτό προσπαθούμε να εργαστούμε. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για το πώς ε, θα ενοποιηθεί αυτό ο τομέας του δικαίου ή πώς θα εναρμονιστεί έτσι ώστε όλες οι δικαιοδοσίες να μπορούσαν να συμφωνήσουν. Το ένα είναι να αναφερθούμε στη Σύμβαση Τρουά του 1995 που θεσπίζει μια σειρά κανόνων που προσπαθούν ε, να ουσιαστικά να βρουν ένα συμβασμό ανάμεσα στις διάφορες νομικές ε, παραδόσεις. Ένα άλλο ε, νομοθέτημα είναι το κοινό πλαίσιο αναφοράς. Προσπαθούμε εκεί να απαντήσουμε στο ίδιο ερώτημα για το πώς ε, θα ρυθμίσουμε την απόκτηση καλή την πίστη λελατημένων έργων τέχνης ή κλεμμένων έργων τέχνης. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ε, πολύ μεγάλη προσταμένη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μία και μόνο νομοθεσία για ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Το δεύτερο θέμα που θίξατε έχει να κάνει με τα λεντυμένα έργα τέχνης από τους Ναζί ή με την ε, απικιακή τέχνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με την ιστορική μας ευθύνη απέναντι στο παρελθόν. Όμως, πέρα από τα κλεμμένα έργα τέχνης από τους Ναζί, Υπάρχει και το θέμα της απικιακής τέχνης, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι, και άλλων εργών ε, που έχουν μεταφερθεί από τα κράτη πηγή σε κράτη εμπορίας και πιο συγκεκριμένα σε κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες ε, από ηθική καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για το επίπεδο ε, των ε, αιτήσεων ε, και το άλλο επίπεδο είναι των ηθικών αποφάσεων. Σε αυτό αναφερθήκαμε σήμερα σε σχέση με τα λελειδημένα έργα τέχνης από τους Ναζί. Ένα τρίτο επίπεδο θα είναι να εισαγάγουμε τέτοιους μηχανισμούς, διαμεσολαβήσεις, διαπραγματεύσεις σε σχέση με την αφρικανική τέχνη, όπως αναφέρατε κι εσείς, αλλά και σε σχέση με άλλες κατηγορίες έργων τέχνης. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλα αυτά τα τρία επίπεδα και να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και στα τρία αυτά επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Φαίνεται ότι εδώ ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις. Απλώς να πω ότι σε ό,τι αφορά τα κλεμμένα έργα τέχνης από τους Ναζί, χάσαμε έναν από τους εταίρους ε, γιατί από την 1η ε, Οκτωβρίου ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Κληρονομιάς ΣΟΑ σταμάτησε να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν πρακτικά έναν λιγότερο συνομιλητή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το σημείο. Ε, θα περάσουμε στο σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων για το συνδυασμό επαγγελματική και δυτικής ζωής, για τους γονείς και τους φροντιστές. Το λόγο έχει η κυρία Μπερζερόν που είναι η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με συγχωρείτε. Γνωμοθετούμε για αυτή την πρόταση οδηγία σε σχέση με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η αρμόδια Επί τη ουσία Επιτροπή είναι Επιτροπή Απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η πρόταση οδηγίοντα καλύπτει την ανάγκη να υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση ω προ την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή, έχοντα υπόψη τι εξελίξει τη κοινωνία τι τελευταίε δεκαετίε κυρίως εδώ αναφέρονται στο θέμα της ε, σύνθεσης ε, των οικογενειών. Το κείμενο προτείνεται από την Κομισιόν ε, θέλει να εξυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην αντιμετωπίση, την εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να τις υποστηρίξει να ακολουθήσουν τη στεδιοδρομία τους και να να συνδυάσουν οικονομική και επαγγελματική ζωή. Έτσι, λοιπόν, τίθεται τα ελάχιστα κριτήρια για ισότητα μεταξύ των δύο φέλων σε ό,τι αφορά τι ευκαιρίε στην αγορά εργασία και τη μεταχείριση στην εργασία. Κανεί δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν μισθολογικέ αποκλήσει αλλά και στι συντάξει μεταξύ των δύο φύλων. Το σημερινό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωση και κρατών μελών έχει λίγες διατάξεις ε, προκειμένου και οι άνδρες να αναλάβουν ε, τις δικές τους ευθύνες στο οικογενειακό επίπεδο έναντι των γυναικών και πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Εγώ προσυπογράφω τις ε, συγκεκριμένους στόχους της πρώτης οδηγίας που θέλει να βελτιώσει την πρόσβαση σε τρόπους που επιτρέπουν τη συμφιλίωση επαγγελματική και ιδιωτική ζωής καθώς και να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις άδειε, τι ε, γονικές άδειε για τους ε, άνδρες. Ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι άνδρες και οι γυναίκες να λαμβάνουν ισότιμα τις γονικές άδειε. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα επειδή υπάρχουν πολύ μικρές αμοιβέ στην περίπτωση της γονικής άδεια, Η πρόταση της Κομισιόν ε, ουσιαστικά να δίνεται, μια, ε, να δίνεται ένας μισθός ε, ανάλογος, η μισή ανάλογη όπως αυτή που γίνεται στην αναρωτική άδεια, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν θέλουμε να προστατεύσουμε το ανώτατο συμφέρον του παιδιού, ε, το οποίο πρέπει ουσιαστικά ισορροπημένα να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς. Πιστεύω λοιπόν ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει ισότιμα να συμμετέχουν στην υποστήριξη της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά το θέμα των ε, μόνων γονέων τίθεται εδώ και εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν προσεγγίζει την κατάσταση ε, ουσιαστικά ελλειπτικά. Ε, ουσιαστικά πρόκειται εδώ για μια πρόταση εξάλληψης ε, των ανισοτήτων ε, των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και την ανατροφή των παιδιών. Η πρόταση οδηγίας ε, αφορά και όσους παρέχουν βοήθεια, δηλαδή ε, τα άτομα που προσφέρουν βοήθεια στην οικογένεια σε μία, ε, σε μία κοινωνία που γυράσκει όλο ένα και περισσότερο. Είναι σημαντικό να προσφέρεται φροντίδα σε ηλικιωμένους ανθρώπους, σε εξαρτημένους ανθρώπους ή σε άτομα με αναπηρία. Ε, παραδείγματο χάρη, χρειάζεται να φροντίζουμε τα γεύματα, τη μεταφορά, την υγιεινή των ανθρώπων αυτών ε, ή μπορεί παραδείγματο χάρη να πρέπει να φροντίζουμε απλώ ε, και για απλά καθήκοντα όπω το να κλείσουν κάποια ραντεβού το να βρούμε μία κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ιδιωτική και επαγγελματική ζωή είναι αναγκαιότητα καθώς δεν είναι λογικό άτομα που έχουν επιλέξει να βοηθήσουν ένα συγγενή να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Η Κομισιόν προβλέπει να βοηθήσει τους φροντιστές στο κείμενό της προκειμένου να συμφιλειώσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Νομίζω παρόλα αυτά ότι μπορούμε να πάμε πιο μακριά από αυτή τη μόνη πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι ένα φροντιστή που έχει σταματήσει τη δουλειά του για να βοηθήσει έναν άπειρο ή ένα άρρωστο παιδί ή έναν άρρωστο θα έπρεπε όχι μόνο να λαμβάνει ένα μισθό γιατί εξοικονομεί χρήματα από το κράτο, αλλά θα έπρεπε να έχει και δικαιώματα συνταξιδότηση. Ε, αρκετά λοιπόν σημεία υπάρχουν σε αυτή την ε, πρόταση οδηγία και υπάρχουν διάφορα στοιχεία που προωθούνται. Θα ήθελα να ακούσω και τι δικέ σα ε, προτάσει για το θέμα αυτό. σα. ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέψετε να συνεχίσω τα αγγλικά διότι ο Σάντο, ο κύριος Γκασπάρ ε, δεν προλαβαίνει να έρθει σήμερα και με παρακάλεσε να διαβάσω ένα σημείωμα που μου έχει δώσει και που περιέχει τη γνωμοδότησή του ή τη γνώμη του τέλος πάντων για τη σημαντική αυτή πρόταση ως ομάδα υποστηρίζουμε την πρόταση νέας οδηγίας που καταργεί την υπαριθμόν 2010-18 και που θα είναι από τα πιο, ε, πιο σημαντικές και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την ισότητα των φύλων και γι' αυτό χρειάζεται από την πολιτική μας ομάδα ε, πολύ προσοχή. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην ζωή πολλών Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών και θα αντιμετωπίσει ελλείψεις σε ε, παροχή φροντίδας, σε ε, εργασιακές ρυθμίσεις, το δικαίωμα αγωνικής άδειας για τους πατεράδες και το καθεξής. Λυπούμεθα που δεν έχουν καταφέρει μετά από την διαδικασία συνδιαλλαγής να καταλήξουν σε συμφωνία, διαδικασία συνδιαλλαγής η οποία κράτησε σχεδόν δύο χρόνια υποστηρίζουμε το αίτημα των συνδικάτων να ζητήσουν επανεξέταση της οδηγίας ή μάλλον αναθεώρηση οδηγίας για τη γονική άδεια και ε, τα σχετικά με τα μισθολογικά. Η σημαντική προτεραιότητα της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είναι μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών για την πρόσβαση στις αγορές εργασίας η απασχολησιμότητα των γυναικών υστερεί τη των ανδρών κατά 12%. Και επειδή ε, αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων μιλών τη οικογένεια, ε, υστερούν. Το συνολικό δε κόστος για την ε, μη δραστηριοποίηση των γυναικών σαν εργατικό δυναμικό είναι της τάξης των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή σημαντικό ποσοστό του ΕΠ. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση νομοθετική για να βελτιωθεί η διαφάνεια και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική οδηγία. Στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα πρέπει να στηριχθούν όλες οι, όλες οι προσπάθειες για την πραγματική εφαρμογή της προτάσεως και ξεκινώντας από τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής. Από τη νομική σκοπιά είναι σημαντικό να τονιστεί στην γνωμοδότηση, να τονιστούν μάλλον όλα τα σημαντικά στοιχεία του νομικού ε, ε, πλαισιού και του πλαισιού πολιτικής για την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής, να υπάρξει νομική βεβαιότητα όπως ζητεί και η μελέτη αντικτύπου. Και τελευταίο σχόλιο του συναδέλφου μου, αναμένουμε ένα ξεκάθαρο ορισμό όλων των μιζώνων προβλημάτων για την εφαρμογή των διαφόρων νομικών πλαισίων, για την εγκυμοσύνη, για την ε, προστασία και κατά των διακριτικών μεταχειρήσεων. Αυτά λέει το σημείο του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Η κυρία Εσταράς Φεραγκούτ. Ευχαριστώ. Πράγματι αυτή η οδηγία αποτελεί μέρος του πακέτου των μέτρων για να υλοποιήσει η Κομισιόν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως προς την εξισορρόπηση επαγγελματική και ιδιωτική ζωής και την βελτίωση της επεκπροσώπησης ε, των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επίσης, ε, θέλει να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που είναι στο 16% και να δοθούν κίνητρα στου άνδρες για να ε, συμφιλιώσουν ε, την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, αλλά να μπορούν και να λαμβάνουν ε, και άδειε, γονικέ άδειε, και να έχουν ευέλικτη μορφή εργασία. Εμείς όλοι συμμεριζόμαστε τους στόχους. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία για να δώσουμε κίνητρα στην άδεια πατρότητας. Η οδηγία θέλει να ενισχύσει λοιπόν αυτή τη γονική άδεια ε, και ουσιαστικά εισάγει και κάποιες διατάξεις ε, που αφορούν ε, τους φροντιστές ατόμων με ειδικέ ανάγκε ή ηλικιωμένων ατόμων. Και συνήθω συνεχίζουν να είναι γυναίκε αυτέ οι φροντιστέ. τώρα, σε σχέση με τι τροπολογίε, εγώ χαιρετίζω όλες ε, τις ε, παραπομπές στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κείμενα. Βεβαίως, η πρωτοβουλία της Κομισιόν στο να δώσει κίνητρα από την πλευρά των ανδρών να παίρνουν άδεια σε πατρότητας είναι κάτι καλό. Και βέβαια θα δούμε και το θέμα ε, των κυρώσεων, πώς θα διαμορφωθεί, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν την οδηγία ε, να ε, μπορούν να τους επιβληθούν κυρώσεις αν δεν εφαρμόζουν την οδηγία αυτή. Πάντως, ε, υποδεχόμαστε θετικά την οδηγία αυτή και νομίζω ότι θα δούμε πώς μπορούμε και να βελτιώσουμε το κείμενο. I do not see any other... Δεν νομίζω να θέλει να πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Δεν βλέπω κάποιον άλλον συνάδελφο. Μήπως θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι στο επίπεδο αυτό καταγράφουμε τα όσα υπόθηκαν. Προς ενημέρωσή σας πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια συνεδρίαση στα πλαίσια του Συμβουλίου με το οποίο συζητούμε και την οδηγία αυτή. Δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες προτού ε, προχωρήσετε κι εσείς περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή στην περαιτέρω ανάλυση της πρότασης αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό. Κανονικά πρέπει να προχωρήσουμε τώρα με τα κοινά σημεία 6, 7, 8 και 9 αλλά δυστυχώς ο εισηγητής μας, ο κύριος Τζαμπάσκι, είναι ακόμα στο αεροπλάνο του. Δεν έχει έρθει ακόμα. Επομένως θα πρέπει να αναβάλουμε την εξέταση των τεσσάρων αυτών σημείων και σας προτείνω, μάλλον το επόμενο σημείο προβλέπεται να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Όσοι λοιπόν δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής ε, στην συνεδρία και κλεισμένο των θυρών παρακαλούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα.